Presidente Knobloch, Πρόεδρε Γκράουμπλοκ, ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μα. Ε, Εξοχότητε, ε, ξέρετε, προσκεκλημένοι μα, ε, πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόεδρε του Ελληνικού Συνεδρίου, κύριε Πρωθυπουργέ, εκπρόσωποι τη Ρουμανικής κυβέρνηση, κύριε και κύριοι, σήμερα εορτάζουμε μια μέρα μνήμης την μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος. Οι κοινότητες των Εβραίων, οι οθνοτικές μειονότητες, όπως η Ρωμά και η Σύντη, όσοι θεωρούνται ανεπιθύμητοι και θεωρήθηκαν ανεπιθύμητοι από το ναζιστικό καθεστώς. Για πρώτη φορά η μέρα μνήμης ε, λαμβάνει χώρα ως τελετή στην, ε, ε, στο εμικύκλιο, στην αίθουσα του εμικυκλίου του Κοινοβουλίου στη Σύνοδο της Ολομέλειας. Με αυτή τη χειρονομία αποστέλουμε ένα ισχυρό μήνυμα περισσότερο από ποτέ. Εμείς δεν ξεχνούμε, δεν ξεχνούμε και δεν θέλουμε να λησμονήσουμε. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη και να καταπολεμήσουμε αοκνός κάθε μορφή μίσους και διακριτικής μεταχείρισης ή αντισημιτισμού. Θέλουμε να παραμείνει ζωντανή η μνήμη των ανίποτων εγκλημάτων του ολοκαυτώματος. Δεν είναι όμως απλώς μία ε, ε, τελετή αυτό. Είναι μια κίνηση για το συλλογικό μας ασυνείδητο, για τη συλλογική μας, τη μας μνήμη. Πρέπει να παραμείνει ένα γεγονό που ποτέ δεν θα ξεχαστεί το όλο καύτωμα. Αυτέ τι πράξει βία και φιλετικού μίσου δεν πρέπει να τι λησμονήσουμε ποτέ. Βάσει των δεδομένων του τελευταίου Ευρωβαρομέτρου, το 50% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί ότι ο αντισημιτισμός είναι ένα πρόβλημα που αφορά την ίδια του τη χώρα. Αυτό καταδεικνύει ότι ο ιός του αντισημιτισμού δεν έχει ακόμη εκριζωθεί. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε με πυγμή και να αντιμετωπίσουμε, ε, να ξεριζώσουμε κάθε σπέρμα μίσους που έχει απομείνει. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη ανεκτικότητας και την βία. Η Ευρώπη έχει ήδη αποδείξει επανειλημμένως ότι μπορεί να το κάνει. Το Ευρωκοινοβούλιο υπήρξε και πάντοτε θα βρίσκεται στο πλευρό όσων είναι θύματα πράξεων μίσου και διακριτική μεταχείρισης. Το 2016 διοργανώσαμε μια σύσκεψη υψηλού επίπεδου για το μέλλον των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Το 2017 εγκρίναμε το πρώτο μας ψήφισμα κατά του αντισημιτισμού. Μαζί από κοινού θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να προασπιστούμε τις αρχές του ε, ψηφίσματος του ΟΗΕ που όρισε μέρα μνήμης τη σημερινή. Θα πρέπει να προωθήσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, να ε, καταπολεμήσουμε οποιαδήποτε άρνηση του ολοκαυτώματος και να καταδικάσουμε χωρίς αντιβολία ε, αμφιβολία κάθε δείγμα διακριτικής μεταχείρισης λόγω εθνοτικής ή θρησκευτικής ε, διαφοράς θα πρέπει ε, να υπάρξει ο σχετικός διάλογος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει χώρος για μίσος και αντισημιτισμό. Δεν θα επιτρέψουμε τα τραγικά σφάλματα του παρελθόντος να επαναληφθούν ποτέ ξανά. Θέλουμε να ακούσουμε την μαρτυρία του Προέδρου Κόρτλοκ, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του Μονάχου. Η Σαρλότ Κόρτλοκ ήταν μόνο τριών όταν της απαγόρεψαν να παίζει με τα άλλα παιδιά στη γειτονιά τη ήταν Εβραία και αυτό ήταν το μόνο της αμάρτημα. Επέζησε όμως από τις φρικαλαιότητες του ολοκαυτώματος χάρη σε μια γυναίκα, μια χριστιανή που ε, δούλευε στην οικογένειά της. Η Σαρλότ Γκλόμποκ ε, αφιέρωσε τη ζωή της στην καταπολέμηση του μίσους και του αντισημιτισμού. Σε εκείνην απευθύνουμε όλοι μας την ευγνωμοσύνη σας ε, προσκαλώ να έρθετε στο Προεδρείο και να λάβετε το λόγο ενώπιον της Συνόδου Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου. Αξιότιμε Πρόεδρε κύριε Ταγιάννη, σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας, τα κατανευναστικά σας ε, λόγια και τα θαυμαστά σας λόγια. Αξιότιμε Πρόεδρε Γιούνκερ, εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Μισελ, ε, αγαπητοί παρόντες μαθητές, ε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμότατα για την πρόσκληση την οποία δέχτηνε με μεγάλη ευχαρίστηση. Διότι για μένα μια επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάντα κάτι το ξεχωριστό. Θέλω να σας πω κάτι ως προσκεκλημένη σε εσά που συνηθίζετε να εργάζεστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πραγματικά ε, ένα ξεχωριστό συνέστημα. Μας δίνει ανάταση ε, το κοινοβούλιο αυτό διαφέρει από όλα τα άλλα. Βέβαια, όλοι σας έχετε εκλεγεί από τη χώρα σας και από το κόμμα σας. Έχετε έρθει εδώ για να κάνετε στη δημοκρατική αρένα πολιτική και να προετοιμάσετε και να διαμορφώσετε ένα καλό μέλλον για τους πολίτες της Ευρώπης. Αλλά δεν σταματούν εδώ όλα αυτά. Πίσω από το Προεδρείο και τούτο εδώ το βήμα δεν βλέπετε μία σημαία, αλλά 28. Και στη μέση έχουμε την ευρωπαϊκή σημαία που συμβολίζει την ιδέα της ενότητας της Ευρώπης. Μία ιδέα στην οποία έχετε υποχρεωθεί να είστε προσιλωμένοι εδώ και το Κοινοβούλιο δεν νομοθετεί μόνο, αλλά δημιουργεί και μια κοινότητα. Εδώ βασίζεται η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, στην ελευθερία, στη δημοκρατία, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο ανοιχτό πνεύμα, στην ανεκτικότητα και ε, την επιθυμία για μια ειρηνική συμβίωση. Αυτά σήμερα είναι αυτονόητα στην Ευρώπη και καθορίζουν την καθημερινότητα, αλλά για μας αυτό δεν ήταν καθόλου προφανές και αυτονόητο και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου εδώ. Όταν ήμουν μικρή, έζησα στο πετσί μου πολύ άγρια τη βαρβαρότητα που δεν ήθελε πια να αναγνωρίσει τίποτα ανθρώπινο και χωρίς ενδιασμούς εξολόθρευε και θανάτωνε. Τότε έχασα σχεδόν τα πάντα, πολλούς από τους αγαπημένους μου, το σπίτι μου και την ε, αρχική μου ε, εμπιστοσύνη και πίστη στον κόσμο και στους ανθρώπους. Για πάνω από μία φορά η ζωή μου σώθηκε από τύχη. Ε, πολλές χρόνια ε, ζούσα σε μια κρυψώνα, με ένα ψευδόνυμο και μια ψευδή ταυτότητα. Γιατί αν ήμουν ο εαυτός μου, αυτό θα σήμαινε σίγουρα τη θανατική μου καταδίκη. Σήμερα μπορώ να βρίσκομαι εδώ ενώπιόν σας, γιατί ε, μεταξύ όλων αυτών των πολλών δολοφόνων, συνοδοιπόρων και παρομοίων, υπήρχαν και άνθρωποι που ρηψοκινδύνευσαν την ίδια τους τη ζωή για να διατηρήσουν την ανθρωπιά τους. Βρίσκομαι εδώ ενώπιό σας, διότι το φως της ανθρωπιάς δεν έσβησε ποτέ εντελώς, ακόμα και στις πιο σκοτεινές εποχές της ανθρώπινης ιστορίας. Αλλά και εδώ είχα καταλάβει από την αρχή με πρώτη ευκαιρία θα έπρεπε να φύγουμε, ο άνδρας μου και εγώ, από την Ευρώπη. Γιατί ε, θεωρούσαμε εκείνη την Ήπειρο διεφθαρμένη και παντού, οπουδήποτε θα ξεκινούσαμε μια νέα ζωή παρά εδώ. Στη συνέχεια γεννήθηκαν τα παιδιά μας και συνεχώς αναβάλαμε την αποδημία μας. Και τα παιδιά μας γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε μια χώρα ε, όπου η αβεβαιότητα και η δυσφορία ε, ήταν τα κυρίαρχα συναισθήματα για εκείνα και για όλη την εβραϊκή κοινότητα. Τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο ε, είχαμε μια αβεβαιότητα. Δεν ξέραμε ε, ποιον έπρεπε να συναστραφούμε που να μην ήταν Εβραίος, γιατί δεν ξέραμε ποιος είχε τα χέρια του αιματοβαμμένα με εβραϊκό αίμα. Και ζούσαμε σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη χώρα ε, να παραμείνουμε στη Γερμανία στο για μας ήταν κάτι το αδιανόητο. Το γεγονός ότι σήμερα βρίσκομαι εδώ ενώπιόν σας είναι ίδια η απόδειξη ότι ευτυχώς κατά τη διάρκεια των δεκαετιών άλλαξαν πολλά και έγιναν πολλά δυνατά τα οποία στο παρελθόν θα θεωρούσαμε αδιανόητα. Ποιος θα είχε άραγε τότε σκεφτεί, υπολογίσει ότι η δημοκρατία μετά τον πόλεμο ε, ε, θα ήταν τόσο ισχυρή. Ποιος θα πίστευε τότε ότι στην Ευρώπη ε, μέσα σε λίγα χρόνια θα μπορούσαν να ξεπεραστούν εχθρότητες αιώνων ολόκληρων. Και ποιος θα το πίστευε ότι μετά ε, από τις ε, φρικαλαιότητες του ολοκαυτώματος, τις αδιανόητες και πάλι θα μπορούσε να ζήσει ένας Εβραίος στην Ευρώπη. Όλα αυτά σήμερα φαίνονται προφανή. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, δεν είναι καθόλου προφανή και τα επιτεύγματα και οι κατακτήσεις δεν είναι πάντα τόσο σταθερά όπως μπορεί να φαίνονται εκ πρώτης όψεως. Και δυστυχώς αυτές τις μέρες αυτό γίνεται πιο σαφές. Η ελεύθερη και δημοκρατική τάξη στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο σήμερα απειλείται περισσότερο από ποτέ. Και εδώ δεν μιλώ για εξωτερικές απειλές ε, σχετικά με τη δική μας συνοχή η ευρωπαϊκή ιδέα, το ευρωπαϊκό ιδεώδες θα μπορούσε να τις αντιμετωπίσει αυτές τις εξωτερικές. Αυτό που με ενισχύει περισσότερο είναι οι έσωθεν ε, επιθέσεις. Ενωμένη στην πολυμορφία μπορεί να είναι η Ευρώπη και στο μέλλον, μόνο ε, εφόσον ξέρει ποιες είναι οι αξίες της και τις θεωρεί ε, σημαντικές για να τις υπερασπίζεται με αυτοπεποίθηση. Αυτό το μέλλον όμως αναγκαστικά συνδέεται με τη γνώση για το παρελθόν. Στις 27 Ιανουαρίου, ε, στην Παγκόσμια ημέρα μνήμης για τα θύματα του ολοκαυτώματος, θυμηθήκαμε τα 6 εκατομμύρια Εβραίων, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από το 1933 μέχρι το 1945 από την ναζιστική Γερμανία η απελευθέρωση του ε, στρατοπέδου συγκέντρωσης Auschwitz στις 27 Ιανουαρίου έγινε πριν από 74 χρόνια. Όλο και λιγότεροι είναι οι επιζώντες που μπορούν να μιλήσουν από το πρώτο χέρι και να πούν ε, πόσα φρικτά έζησαν εκεί. Γι' αυτό και είναι πιο σημαντικό ε, και περισσότερο σημαντικό το μήνυμα των επικεφαλής των ψηφοδελτίων ε, των χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών για τις επόμενες ευρωεκλογές. Ήταν μαζί ο Μάνφρετ Βέμπερ και ο Φραντ Τίμερμανς στο Auschwitz. Παρ' όλα αυτά παραμένει ένα θλιβερό γεγονός. Όλο και περισσότερο χάνονται αυτές οι φωνές, σβήνουν. Θα έχουμε σε λίγο ένα διάστημα και ένα χρόνο χωρίς αυτόπτες μάρτυρες. Και ορισμένοι θεωρούν ότι δεν χρειάζεται πια να θυμόμαστε ε, αυτά τα πράγματα, το ολοκαύτωμα. Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο λανθασμένο. Παντού βλέπουμε στην Ευρώπη πολιτικά κινήματα, κερδίζουν και δύναμη, τα οποία αποφασισμένα ε, αντιστέκονται στη μνήμη ε, και στις επαιτίους. Προπαγανδίζουν ένα παρόν χωρίς παρελθόν, ως ένα εφαλτήριο σε ένα μέλλον χωρίς μνήμη. Ε, έτσι, με τέτοια λύθη της ιστορίας σηκώνει κεφάλι ο αντισημιτισμός και δυστυχώς αυτό δεν είναι απορίας άξιο Ε, εμείς, τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας, ήδη από σήμερα ζούμε αυτές τις επιπτώσεις και στη Γερμανία και σε πολλά άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να είσαι Εβραίος και να έχεις δημόσια ζωή απαιτεί ε, αστυνομική προστασία ε, και οι Εβραίοι όλο και περισσότερο αισθάνονται ανασφαλείς. Βέβαια γυρίσανε ε, στο κέντρο των πόλων και συναγωγές χτίζονται και σπίτια και αιστείες κοινοτικέ. Είναι μια νέα μορφή συνύπαρξης. Τα κτίρια αυτά βασίζονται στα θεμέλια της εμπιστοσύνης. Και εγώ μπορώ να σας πω από πρώτο χέρι πόσο χρειάστηκε μέχρι να ε, αισθανθώ ε, ξανά μετά το 1945 πόλη μου το Μόναχο που έχω γεννηθεί και είναι η πατρίδα μου. Πραγματικά ε, άδειασα τις βαλίτσες μου με την, τα γένεια της συναγωγής καινούρια στο Νοέμβριο του 2006, οριστικά. Και σήμερα καταλαβαίνω ότι μήπως βιάστηκα να αδειάσω αυτές τις βαλίτσες. Σε ε, πολλές περιπτώσεις αμφιβάλλει ε, ο Εβραίος για το μέλλον του. Οι Εβραίοι πίστευαν ότι ποτέ δεν θα αισθανθούν στη χώρα τους τέτοια πίεση. Είναι πολλές οι επιθέσεις και λεκτικές, αλλά ακόμα περισσότερη η αδιαφορία, η έλλειψη κατανόησης, η έλλειψη ενσυναίσθησης. Γιατί όπου και να γυρίσουμε ε, τη ματιά μας, σηκώνει το άσχημο κεφάλι του ο αντισημιτισμός σε ε, όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε όλο το πολιτικό φάσμα. Δεν είναι μόνο οι ακραίοι, είναι και το κέντρο και πολλοί ε, ε, μουσουλμάνοι. Η AFD, οι BDS και ακραίοι ε, Ισλαμιστές έχουν κοινά. Λίγα κοινά, αλλά στον αντισημιτισμό έχουν κάτι που τους ενώνει όλους. Αξιότιμοι παρόντες. Βέβαια όλα αυτά είναι η μισή αλήθεια και μόνο. Ευτυχώς παντού στην Ευρώπη υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται για τη μνήμη και τη δημοκρατία και την ε, ανοιχτή σκέψη. Οι φωνές τους είναι πολλές, είναι ηχηρές. Σε πολλά, αν όχι σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, συνιστούν την ευρία πλειονότητα του πληθυσμού. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε λόγω αυτής της αριθμητικής υπεροχής. Η ε, ιστορία έχει αποδείξει πόσο δύσκολο μπορεί να είναι το έργο της ε, πλειονότητας όταν θέλει να υπερασπιστεί τα ιδανικά της ε, σε ε, μια επίμονη μειοψηφία απέναντι. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα στην ευρωπαϊκή πολιτική, πόσο γρήγορα διαδίδεται ο αντισημιτισμός εάν δεν μπουν κάποια όρια εγκαίρως. Ένα από τα πιο δραστικά παραδείγματα αυτής της εξέλιξης διεξάγεται σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Εργατικό Κόμμα που κατά τη μακρά της ιστορία ήταν ένα προπύργιο ε, λογικής, της πολιτικής, με την προεδρία του Τζέρεμι Κόρβιν τα τελευταία χρόνια ε, έγινε από το πια κατάφορα προβληματικά κόμματα στην Ευρώπη ε, σε ό,τι αφορά τον πολιτικό αντισημιτισμό. Με τη νέα ηγεσία το εργατικό κόμμα άφησε πίσω του και πολύ μακριά το πολιτικό κέντρο. Είναι προφανές ότι στο ηθικό ημίφος το να μην παίρνει θέση βοηθάει να αναπτυχθούν τα πιο άγρια ζυζάνια της πολιτικής. Πόσο γρήγορα φεύγουμε από την πολιτική της ανοχής και της ανεκτικότητας όταν ε, είναι ευνοϊκά τα σημεία των καιρών. Παράδειγμα λοιπόν είναι το εργατικό κόμμα υπό τον Κόρμπιν και τέτοιες ε, εξελίξεις δεν αφορούν μόνο ε, τον ιδιαίτερο ρόλο του Μεγάλου ε, Ηνωμένου Βασιλείου συγγνώμη, φαίνονται παντού στην Ευρώπη. Κάτι έχει ολιστήσει, κάτι έχει αλλάξει. Ο αντισημιτισμός σε πολλές χώρες της Ευρώπης βρίσκει χώρο και πολιτικό και κοινωνικό ξανά. Ε, αυτό που και πολύ καιρό έρχεται στην επιφάνεια και όπου ο αντισημιτισμός δεν πατάσεται ενεργά και αμέσως ανοίγει δρόμους και το είδαμε πρόσφατα, το είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι παρόντες. Θα ήθελα να είμαι απολύτως ξεκάθαρη. Σε μια Ευρώπη όπου πάνω από το 89% του εβραϊκού πληθυσμού ε, διαμαρτύρεται για την αύξηση του αντισημιτισμού στη χώρα του, ε, είναι προβληματική αυτή η Ευρώπη. Μια Ευρώπη που πάνω από το 1 τρίτο των Εβραίων έχουν σκεφτεί σοβαρά να αποδημήσουν. Έχει πρόβλημα ο αντισημιτισμός δηλητηριάζει γενικά το κλίμα στην κοινωνία. Ελευθερία και ασφάλεια ισχύουν για κάθε πολίτη της Ευρώπης ή για κανέναν. Ο αντισημιτισμός τα περιφρονεί αυτά. Με γεμίζει πόνο και λύπη τόσα πολλά χρόνια μετά το τέλος του ολοκαυτώματος σήμερα να έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τόσο πολύ δεδομένο αντισημιτισμό. Αλλά χρέος όλων μας θα πρέπει να είναι να αντιταχτούμε και να αντισταθούμε σε αυτή την ε, εξέλιξη και να την κάνουμε να υποχωρήσει. Αυτό είναι το δικό μας καθήκον. Διότι η μεγαλύτερη τραγωδία ε, της εβραϊκής ιστορίας έγινε εδώ στην Ευρώπη. Οι πόλεις που είναι σήμερα το κέντρο της ζωής μας, πριν από 80 χρόνια και λιγότερα, ήταν τα θέατρα ε, του χειρότερου εγκλήματος στην ιστορία της ανθρωπότητας και τα προκάλεσε η τότε γερμανική κυβέρνηση. Αξιότιμοι παρόντες, αξιότιμοι επίτροποι, αξιότιμοι βουλευτές. Εσείς είστε εκείνοι που ορίζετε τις μοίρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, γι' αυτό απευθύνω έκκληση σε εσά και σήμερα και στο μέλλον και μετά τις ε, ερχόμενες ευρωεκλογέ να αντισταθείτε ε, στεναρά σε αυτόν τον αντισημιτισμό. Επιθυμώ τούτο το κοινοβούλιο και στο μέλλον να εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στο χρέος που έχει και στην ευθύνη του. Η ελευθερία και η δημοκρατία που απολαμβάνουμε σήμερα είναι πάντα μόνο τόσο ισχυρή όσο ισχυρή είναι η δέσμευση της δημοκρατίας και των δημοκρατών. Και θα πρέπει η πλειονότητα να αντισταθεί στη μειονότητα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να κερδίσει αυτό το μίσος. Όχι πια, όχι ξανά από το, όχι, το ποτέ πια δεν επιτρέπεται να γίνει και τώρα ξανά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σα ευχαριστούμε εξ ονόματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστούμε για γνώμη για την τόσο πολύτιμη κατάθεσή σα που για μα έχει ανεκτιμητή αξία. Τώρα θα τηρηθεί ενό λεπτού σιγή στην μνήμη όλων των θυμάτων του ολοκαυτώματο. και έχουμε κατά νου το ότι ένα λεπτό για κάθε θύμα θα σήμαινε ότι θα πρέπει να κάτσουμε για πέραν από 11 έτη στην ε, σιωπή. Κατόπιν. Κατά, αυτή, κατά αυτό το λεπτό θα έχουμε προβολή κάποιων σχεδίων ε, παιδικών. Ήταν 15.000 και σώθηκαν 150 και μας ε, άφησαν αυτές τις ε, εντυπώσεις, αυτά τα παιδιά που χάθηκαν με τις εντυπώσεις τους, επομένως και πρόκειται, αυτά έχουν έρθει από την συναγωγή της ε, Πράγας. Εκεί αποτυπώνονται τα συναισθήματά τους ενώπιον αυτών των φρικαλαιοτήτων που κανένα παιδί δεν θα πρέπει πια να υποστεί. Ποτέ πια.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

La seduta è sospesa Διακόπτεται η συνοδός για 5 λεπτά.